Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στη συνέντευξη τύπου. Ευχαριστώ ε, για την παρουσία των διερμηνέων. Επειδή έπρεπε να έχουμε παρουσία των διερμηνέων να αργήσαμε ένα τέταρτο να ξεκινήσουμε, θα μιλήσουμε για τις εκλογές στη Βολιβία και τις, ε, τα συμπεράσματα της ε, αποστολής των παρατηρητών. Ο Χαβιέ έχει το λόγο. Καλημέρα σας. Θα σας πούμε λοιπόν λίγα πράγματα ε, για το τι κάναμε στη Βολιβία στις τελευταίες εκλογές. Ε, μεταβήκαμε εκεί κατόπιν προσκλήσεως ε, των Βολιβιανών εκλογικών αρχών με στόχο την παρατήρηση των γενικών εκλογών της 12 Οκτωβρίου 2014 η αντιπροσωπεία που την ομάδα μας απαρτιζόταν από τη Σοφία ε, Σακοράφη και από τον Χαβιέρ Κάουσα, τον υποφαινόμενο. Και εστιάσαμε κυρίως ε, στην άσκηση ε, του πολιτικού δικαιώματος, ε, της ε, ψήφου δηλαδή, καθολικής άμεσης ψηφοφορίας. Σημειώσαμε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις και τις ανησυχίες για το κατά πόσον ήταν ιδανικές οι συνθήκες ε, συμμετοχή των εκλογών και εκπροσώπησης όλων των ε, πολιτικών ομάδων. Υπήρξαν κάποια παράπονα, αλλά η αποστολή παρατήρησης ε, δεν επιβεβαίωσε ότι αυτές οι καταγγελίες ή τα παράπονα ευσταθούσαν. Αντιθέτως, θεωρούμε ότι υπήρξε πολυφωνία στην εκλογική αντιπαράτευση. Διανεργήθηκαν πολύ σωστά, πιστεύουμε, οι εκλογές είναι πάρα πολύ σωστό ε, και καλό το εργαλείο το οποίο εφαρμόστηκε για ε, να εφαρμοστεί με το βιομετρικό αυτό χαρακτήρα ε, η ταυτότητα όλων των εκλογέων. Αυτά τα ψηφοδέλτια, μάλλον πώς να το πω, ήταν υπογεγραμμένα από τρία άτομα, υπήρχαν και δακτυλικά αποτυπώματα. Άρα και ακόμη και το, το, είδος των ψηφοδελτίων μας δίνει εγγύησεις στις 12 Οκτωβρίου λοιπόν έγιναν εκλογές ε, οι οποίες πληρούσαν όλες τις διεθνείς ε, προδιαγραφές και συμφωνίες, ήταν δίκαιε, ήταν διαφανείς. Επιβεβαιώσαμε επί ότι η εκλογική εκστρατεία, η προεκλογική εκστρατεία έγινε απόλυτα ομαλά φυσιολογικά. Ε, επισκεφθήκαμε και τα εκλογικά τμήματα και μπορεί να σας δώσει λεπτομέρειες η Σοφία στη συνέχεια για το τι κάναμε εκεί, ποια ήταν η δράση μας και όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων ε, και στην αντιπολίτευση όλοι συμφώνησαν και υπέγραψαν για το ότι οι εκλογές διεξήχθησαν ε, απόλυτα ε, κανονικά και φυσιολογικά. Υπήρχε μυστική ψηφοφορία και είχε και νόημα να γίνει έτσι αλλά υπήρξε επίσης και δυνατότητα να παρασχεθεί συνδρομή σε όσους δεν μπορούσαν να ψηφίσουν από μόνοι τους ε, και υπήρχε και σε μπράγ ε, το ψηφοδέλτιο δηλαδή για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Είδαμε λοιπόν επισκεφτόμενοι δειγματοληπτικά κάποια εκλογικά τμήματα ότι όλα πήγαν ε, καλά. Υπήρξε απόλυτη ηρεμία, επικράτησαν τα, τα ήρεμα πνεύματα. Θα σας πω τώρα για τις κάποια άλλα θετικά, η συμμετοχή ε, στις εκλογές ε, και ως εκπρόσωποι, δηλαδή και στο εκλέγει και στο εκλέγεστε, ενώ γυναικεία εκπροσώπηση, μας φαίνεται ε, σημαντικό να πούμε ότι προστατεύονται ιδιαίτερα οι γυναίκε με τον εκλογικό νόμο 243 κατά της παρενόχλησης και της άσκηση κατά των γυναικών οποιοδήποτε υποψήφιος ε, διώκεται για ε, βία, ε, αρσενική βία κατά γυναίκας δεν μπορεί να συμμετέχει στις εκλογές. Και επίσης και οι αυτόχθονες προστατεύονται, υπάρχουν ειδικέ διατάξεις με την νομοθεσία αυτή, αυτό το εκλογικό νόμο δηλαδή που πραγματικά εγγυάται τον πολυφωνικό, πλουραλιστικό χαρακτήρα του βολιβιανού κράτους. Επίσης, ε, ξέρετε ότι η γεωγραφική κατάσταση στη χώρα είναι κάπως ιδιόμορφη, είναι ιδιαίτερη ε, και υπήρχαν ε, κάποια στοιχεία γεωστατικά. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν εξοπλισμένα με την κατάλληλη τεχνολογία. Επίσης τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούσαν να ψηφίσουν, όπως είπα υπήρχε συνδρομή, είτε συνοδεύονταν είτε δεν συνοδεύονταν, πάντα όμως υπήρχε ένας μάρτυρας ε, και έπειτα ε, είδαμε ότι υπήρχε και στις διάφορες ε, γλώσσες των αυτοχθόνων στις γλώσσες τους υπήρχε ενημέρωση, είδαμε τα έγγραφα, υπήρχε και ένα πρόγραμμα για την νεολαία που ενημέρωνε και βοηθούσε τους νέους να ψηφίσουν, τους νεαρούς ψηφοφόρους και είδαμε πολύ μεγάλη διαφάνεια. Ήταν σαν όλη η να είναι μια κάλπη. Διότι το ανώτατο εκλογικό δικαστήριο κάλεσε πολλούς ε, πολλές αποστολές κάλεσε εμάς, έτσι, αλλά και από τον ΟΗΕ, την Ουνασούρ, τη Μερκοσούρ, το Παρλαθέν, ε, κάλεσε από, τις, ε, από την κοινωνία των πολιτών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι υπήρξε οποιαδήποτε μεροληψία. Επίσης, ε, αντίθετα με το ότι συμβαίνει στην Ευρώπη, αυτό το δικαστήριο, το εκλογικό, είναι ανεξάρτητη αρχή, ανεξάρτητη εξουσία στη Βολιβία και εγγυάται την ανεξαρτησία. Τώρα, υπήρξαν κάποιες αρνητικές πτυχές ε, Είδαμε ότι υπήρξαν κάποια φυλάδια προπαγάνδας εκλογικής τα οποία είχαν ρίξει κάποια από τα εκλογικά τμήματα. Κάποια εκλογικά τμήματα δεν ήταν εύκολα προσβάσιμα επίσης. Επισκεφθήκαμε και ένα σοφρονιστικό κέντρο και είδαμε ότι ήταν δύσκολο οι τρόφιμες ε, ε, των φυλακών να μπορούν να ψηφίσουν. Ήταν λίγο δύσκολο και ζητήθηκε να υπάρξει συντονισμό του ε, εκλογικού δικαστηρίου για να μην καταδικαστεί διπλά αυτό το άτομο είναι τρόφιμο φυλακών ενό οπνευστικού ιδρύματο, αλλά έχει παρόλα αυτό το δικαίωμα να ψηφίσει. Δεν μπορεί να τιμωρηθεί διπλά. Επίση, είδαμε ε, κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά την μηχανοργάνωση, ε, αν μπορούσε δηλαδή ε, σε περίπτωση αμφιβολίας να βοηθηθεί κανείς με, το, με τα κομπιούτερ. Βέβαια ήταν ελάσσονα προβλήματα αυτά ε, οργανωτικά και σε καμία περίπτωση δεν υπονομεύουν το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης όπως είπα υπήρχε ελευθερία, υπήρχε πολυφωνία, το είδαμε, το βιώσαμε, μας κάλεσαν σε σταθμούς τηλεοπτικούς και επισκεφθήκαμε διαφόρων τάσεων ε, μέσα ενημέρωσης. Και εκεί βιώσαμε πραγματικά ότι ακούστηκαν ε, πολλές και διαφορετικές απόψεις και εκφράστηκαν όλες αυτές από τα μέσα επικοινωνίας. Και θεωρούμε επίσης ότι τηρήθηκαν ε, και τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές ε, όταν υπήρχε προσβολή κάποιες υποψηφιότητας και έπρεπε να συζητηθεί το κατά θεωρούμε ότι είναι υψηλός ο βαθμός ε, ε, ε, του εκδημοκρατισμού, αν θέλετε, της, του δημοκρατικού χαρακτήρα της βολιβιανής κοινωνίας και θα δώσω τώρα το λόγο στη Σοφία. Λοιπόν, να σας καλημερίσω, να ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Κινδυνεύοντας να επαναλάβω βεβαίως τα όσα είπε ο, ο Χαβιέ, αλλά θα είναι σαν επιβεβαίωση και της παρουσίας μας, αλλά κυρίως του γεγονότος ότι είδαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα και δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην, στην έκθεση που θα παρουσιάσουμε. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ επιγραμματικά σε διαδικαστικά θέματα και αν έχουμε χρόνο θα κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό που πιστεύω ότι συμβαίνει σήμερα στη Βολιβία. Ε, σαν αποστολή φτάσαμε στη Βολιβία το βράδυ της 9ης Οκτωβρίου. Οι εκλογές εκεί διεξάγονται από ανεξάρτητη αρχή που δεν έχει καμιά διασύνδεση με το κράτος και αυτό το αναγνωρίζουν και το σέβονται όλοι, κυβέρνηση, αντιπολίτευση και ψηφοφόροι. Η ψήφο προβλέπεται στο Σύνταγμα υποχρεωτική, με μόνε κυρώσει, την επιτρίμηνα απαγόρευση τραπεζικών συναλλαγών και την έξοδο από τη χώρα. Σε αυτέ τι εκλογέ ψήφισαν και οι νέοι από 18 χρονών. Οι εκλογικοί κατάλογοι για πρώτη φορά περιελάμβαναν και βιομετρικά χαρακτηριστικά, όπω είπε και ο Χαβιέ, δηλαδή φωτογραφία, οικογενειακή κατάσταση κλπ. Σε όσες περιοχές χρειαζόταν τόσο το ενημερωτικό υλικό όσο και τα ψηφοδέλτια ήταν γραμμένα στις τοπικές διαλέκτους και αυτό εξαιτίας του πολυεθνωτικού ε, πεδίου που υπάρχει στην, στην περιοχή. Περίπου ήταν σε τέσσερις διαλέκτους. Την Παρασκευή λοιπόν στις 10 Οκτωβρίου κάναμε συναντήσεις ε, με τα μέλη των διεθνών εκλογικών αποστολών, των παρατηρητών και είχαμε ενημέρωση για όλη την διαδικασία από την ανεξάρτητη αρχή της προετοιμασίας και της διεξαγωγής των εκλογών. Συναντηθήκαμε με υποψηφίους και εκπροσώπους τους από όλα τα κόμματα για την Προεδρία, Αντιπροεδρία, Γερουσία, Βουλή, Αντιπροσώπων και εκπροσώπους σε υπερεθνικούς οργανισμούς του κράτους της Βολιβίας. Στη συνάντηση αυτή η αποστολή της GUNGL κατέγραψε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που αναφέρθηκαν από διάφορους παράγοντες. Συγκεκριμένα σε αυτές τις συναντήσεις εκφράστηκαν και ανησυχίες για την επάρκεια των δυνατοτήτων της εκλογικής αρχής, την ακρίβεια και την αξιοπιστία των εκλογικών καταλόγων και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εκλογές από διάφορες δυνάμεις. Ειδικότερα μας εκφράσαν υπόνοιες για πιέσεις από την κυβέρνηση ως προς την ψήφο των δημοσίων υπαλλήλων, Επίσης εκφράστηκαν και παρατηρήσεις για τη συμπεριφορά της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Την Κυριακή, από τις 7 έως και τις 3, κάναμε επισκέψεις στα παρακάτω κτίρια που φιλοξενούσαν εκλογικά κέντρα, όπως ε, γυναικείες φυλακές του Μυραφλόρες, το Τεχνολογικό Κολέγιο του Αγιακούχο και το Κολέγιο Αβε Μαρία, το Κολέγιο Καστίγιο. Στα κτίρια αυτά συναντήσαμε και συνομιλήσαμε με τις ευθορευτικές επιτροπές περίπου 75 διαφορετικών εκλογικών κέντρων. Από τις 3 μέχρι τις 6 πήγαμε στο κολέγιο Λαπάς. Σε αυτό το κτίριο παρακολουθήσαμε το κλείσιμο των καλπών, την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και την τελική καταγραφή των αποτελεσμάτων σε 6 διαφορετικά εκλογικά κέντρα. Τα μέλη της αντιπροσωπείας είχαν απόλυτη ελευθερία κινήσεων και επαφών κατά την επίσκεψή τους στα εκλογικά κέντρα συζήτησαν με πάρα πολλούς ψηφοφόρους, με πάρα πολλά μέλη των εφορευτικών επιτροπών και κυρίως με πάρα πολλούς διαφορετικούς εκπροσώπους όλων των κομμάτων που ήταν παρατηρητές των εκλογών. Σε καμιά περίπτωση δεν καταγγέλθηκε στα μέλη της αντιπροσωπείας κάποιο σοβαρό παράπτωμα ή πρόβλημα για τη διαδικασία. Η εξυπηρέτηση όσων δεν γνώριζαν που ψηφίζουν ή δεν έβρισκαν το όνομά τους στις λίστες μπορούμε να πούμε ότι ήταν σχεδόν πλήρης. Επίσης, η εξυπηρέτηση όσων ψηφοφόρων δυσκολεύονταν να φτάσουν στην κάλπη, όπως ανέφερε και ο Χαβιέ, κυρίως των ηλικιωμένων, ήταν άρτια. Ιδιαίτερα πρέπει να σημειωθεί ότι η πρόνοια για δεν μπορούσαν να μεταβούν στα εκλογικά κέντρα, άρρωστοι, ανάπηροι, λεχόνες κλπ, καθώς και η διαθεσιμότητα του συστήματος Μπράι. Υπήρχε ειδική οργάνωση, η οποία είχε καταγράψει την πλειοψηφία των περιπτώσεων και αντιμετώπισε με επιτυχία και τις περιπτώσεις που προέκυψαν την ημέρα των εκλογών. Όλα τα παραπάνω συνέτειναν ώστε η γενική ατμόσφαιρα που επικράτησε όλη την ημέρα των εκλογών να είναι ομαλή και ειρηνική σύμφωνα με τα όσα παρατήρησε και διαπίστωσε η αντιπροσωπεία μας για το τι συνέβη την ημέρα των εκλογών, δεν επιβεβαίωσε ούτε στο ελάχιστο το βάσιμο των παρατηρήσεων και των επιφυλάξεων που είχαν εκφραστεί, καθώς δεν βρήκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να τα τεκμηριώνει. Εδώ πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνήμα για τη δυνατότητα που δόθηκε για πρώτη φορά σε Βολιβιανούς, υπήκοους, κατοίκους εξωτερικού να ψηφίσουν, εκ των οποίων ψήφισαν περίπου οι 160.000. Κατά τη συνολική εκτίμησή μας, οι εκλογές της Κυριακής 12 Οκτωβρίου έγιναν σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα για δίκαιες εκλογές. Η μέρα των εκλογών εξελίχθηκε ομαλά στα διαφορετικά εκλογικά τμήματα που επισκεφθήκαμε, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από όλα τα αντίπαλα μέρη. Πιστεύουμε ότι πρέπει να συγχαρούμε πρώτα και κύρια το λαό της Βολιβίας για τη μαζική συμμετοχή του στις εκλογές καθώς επίσης και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό το άρτιο αποτέλεσμα από το απλό μέρος της Εφορευτικής Επιτροπής μέχρι, τον, μέχρι την πρόεδρο της Ανεξάρτητης Επιτροπής της Προετοιμασίας και της Διενέργειας των Εκλογών. Θα μου επιτρέψετε τώρα να πω και δύο λόγια του τι πιστεύω εγώ ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βολιβία. Η Βολιβία αναφέρεται στην επίσημη και πλήρη ονομασία της σαν πολυεθνωτικό κράτος. Αυτό εφαρμόζεται στην πράξη με έναν τρόπο απλό και πολύ ουσιαστικό. Αυτό σημαίνει πλήρη σεβασμό σε εθνοτικές ομάδες του πληθυσμού όσον αφορά στη γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμά τους, θρησκεία και τις λατευτικές τους εκδηλώσεις και την απρόσκοπτη και ισότιμη συμμετοχή τους και την εκπροσώπησή τους στις εκλογές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι τα ψηφοδέλτια και οι οδηγίε για την εκλογική διαδικασία, όπω σα είπα και προηγουμένω, είχαν συνταχθεί και σε άλλε γλώσσε και όχι μόνο στα Ισπανικά. η περιγραφή για μένα είναι πάρα πολύ επιγραμματική και αξίζει να αναφερθούμε κάποια στιγμή πιο αναλυτικά γιατί τηρουμένων των αναλογιών και όλων των ιδιαίτερων παραμέτρων που μπορεί να ισχύουν στην Ευρώπη και όχι μόνο, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να διδαχθούμε για την αντιμετώπιση προβλημάτων αυτών που στην Ευρώπη ονομάζουμε μειονότητες, θρησκευτικέ, εθνικές, πολιτισμικές κλπ. Το δεύτερο που θα μου επιτρέψετε να τονίσω είναι η αίσθηση που αποκόμισα για, για το πώς αντιλαμβάνονται τη δημοκρατία οι πολίτες της Βολιβίας. Είναι μια ιδιαίτερη αντίληψη που ξεφεύγει από την κουλτούρα μας και η οποία εμένα μου δημιούργησε την αίσθηση ότι η συνειδητοποίηση του τι έχουν κατακτήσει εκφράζεται και πάλι με έναν εντυπωσιακά απλό τρόπο ότι αυτό είναι κτήμα τους και το υπερασπίζονται θεωρώντας αδιαπραγμάτευτα στοιχεία όπως η διαφάνεια, ο απόλυτος σεβασμός, το απρόβλητο των κανόνων της διαδικασίας και αυτά τα υπερασπίζονται με τη δική του συμπεριφορά. Όπως σας είπα, επισκεφτήκαμε πάρα πολλά εκλογικά κέντρα και αυτό μας το, μας το επιβεβαίωσε. Ε, δεν θα σας αναφέρω για το απλό των εκλογικών ε, ε καλπών, το οποίο εάν το βλέπατε θα σας έδινε την εντύπωση ότι μάλλον είναι ανασφαλές, αλλά επί της ουσίας είχε την απόλυτη ασφάλεια και διαφάνεια, όπως και ο τρόπος που άνοιξαν οι κάλπες και ε, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, όχι μόνο στην Εφορευτική Επιτροπή, όχι μόνο στους υπεύθυνους των κομμάτων οι οποίοι μπορούσαν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, αλλά είχαν δικαίωμα και οι πολίτες να είναι παρόντες στην καταμέτρηση των ε, ψηφοδελτίων. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα επισημάνουμε ε, και να τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας και τα, εμείς τα έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη μας στην έκθεση που θα καταθέσουμε. Κλείνοντας θέλω να μεταφέρω την πεποίθησή μου ότι η ε, επανεκλογή με αυτόν τον πανηγυρικό τρόπο του Ιβο Μοράλες στην Προεδρία για τρίτη συνεχόμενη φορά δεν αφορά μόνο στην ιδιαίτερη προσωπικότητα του Προέδρου αλλά αντανακλά ένα ιδιαίτερο και ιδιόμορφο πείσμα του βολιβιανού λαού να υπερασπιστεί αλλά και να προαγάγει αυτά που μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη αν σας ταλαιπώρησα λίγο παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σακοράφα, σε... η οποία θα εκλεγεί σε μερικές ώρες πρόεδρος της Επιτροπής για τις σχέσεις με την Λατινική Αμερική και πρέπει να πω ότι, ότι ο κύριος Κάουσου είναι αντιπρόεδρος της ΑΦΕΤ. Ε, υπάρχουν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους παρακαλώ. Eh, eh, λοιπόν, σας έστειλα ένα χαρτί με την ερώτησή μου που αφορά εάν όντως μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις ελευθερίας, διαφάνειας, πολυφωνίας. Μπορείτε να μας ε, διαβεβαιώσετε ότι είναι πλήρως δημοκρατικές και πώς εκτιμάτε τη σημασία του ρόλου του Εύω Μοράλες σε αυτή την ε, προεκλογική διαδικασία η χαρισματική ηγεσία του μπορεί να δημιουργήσει κάποιες, κάποιες υποψίες για το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι και στην έκθεση και στις ομιλίες μας καταστήσαμε σαφές ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τη διαφάνεια αυτών των εκλογών. Και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούν και όλες οι άλλες αποστολές παρατήρησης. Σε όλες τις ε, προκαταρκτικές εκθέσεις βλέπουμε ότι ότι το βράδυ όταν οι περισσότερες ε, αποστολές μίλησαν στα μέσα ενημέρωση συμφωνούσαν όλες. Και η τελική μας έκθεση αυτό λέει. Διαπιστώνουμε την πολυφωνία και για την ενημέρωση. Τώρα, τώρα δεν θα πρέπει νομίζω εμείς να αρχίσουμε να εκτιμάμε τι εκπροσωπεί ο, ο Εύω Μολάρης. Αλλά εμένα με κουράζει το ότι ορισμένες φορές κατηγορείται το ότι ε, κάποιος μπορεί να είναι υποψήφιος μία, δύο, τρεις φορές, ενώ στη χώρα μου δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Και ότι όσο ψηφίζονται, τότε επανεκλέγονται. Γιατί εφαρμόζεται αυτό για τον Εύω Μοράλες και άλλες χώρες του Νότου. Ο Φελίπη Κονθάλεθ ε, εξελέγει τρεις φορές. Κανείς δεν το κατηγόρησε ότι ήθελε να μείνει αιωνίως. Εξηγήστε μου τι σημαίνει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να καταγγελθεί αυτό. Δεν είναι ε, εσαή η εκλογή του, είναι με βάση τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Εγώ δεν θέλω τώρα να κάνω ερμηνεία προθέσεων του Εύω Μοράλες, αλλά θέλω να καταγγείλω αυτή τη στρεβλή νέο απικιακή αντιμετώπιση των χωρών, ε, των χωρών του Νότου και ιδιαίτερα αυτών που δεν τα πάνε καλά με τη Δύση. ερώτημα θα, θα, μάλλον θα μπορούσα να απαντήσω πιθανόν στο ερώτημα ε, το γιατί επανεξελέγει, αυτό ρωτάτε, ή υπάρχει αμφισβήτηση για την επανεκλογή του. Γιατί αμφισβήτηση για την επανεκλογή του, αν μου επιτρέπετε να κάνω αυτό το, το σχόλιο, δεν υπάρχει από τη στιγμή που το ποσοστό είναι αυτό που είναι και από τη, τη στιγμή που ο Βολιβιανός λαός επέλεξε τον Ιβο Μοράλες αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή για πρόεδρο του. Euh, est-ce Άλλες ερωτήσεις. Παρακαλώ. Οπωσδήποτε. Σίγουρα σε διάφορες χώρες και εντός και εκτός της Ένωσης υπάρχει δυνατότητα επανεκλογής απεριόριστα. Ωστόσο, κάποιοι θα μπορούσαν να σκεφτούν ότι οι θεσμοί των χωρών της Ένωσης είναι πιο ισχυροί και αντέχουν το ενδεχόμενο να παραμένει ο ίδιος Πρωθυπουργό σε μια χώρα. θεωρείται ότι η Βολιβία είναι θεσμικά έτοιμη για να έχει ένα πρόεδρο, τον ίδιο πρόεδρο, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να πέσει σε καταστάσεις προσωποπαγών καθεστώτων. Απάντηση. Κοιτάξτε. Εμείς διαπιστώσαμε πλήρη δημοκρατία και μάλιστα προηγμένη. Άρα γιατί να μην αποφασίζουν οι ψηφοφόροι ποιος θα είναι πρόεδρος. Γιατί να έχει κάποιος λαός λιγότερες δυνατότητες ε, από άλλους. Είτε όλοι τα κανένας που λέγει το τραγούδι. Γι' αυτό κατηγόρησα αυτήν την στρεβλή απικιοκρατική προσέγγιση. Διότι Διαπιστώσαμε πόσο ισχυρή είναι η δημοκρατική θεσμή στη Βολιβία. Το εξετάσαμε, το, διαπιστώσαμε. Και το ανώτατο εκλογικό δικαστήριο κάλεσε διάφορες ε, αποστολές παρατηρητών, είχαμε κάθε ελευθερία να ρωτήσουμε όποιον θέλουμε, να πάμε όπου θέλουμε, να μιλήσουμε με στρατιωτικούς, με ε, αστυνομικούς των ειδικών δυνάμεων, με κοινούς αστυνομικούς και διαπιστώσαμε ότι υπήρχε και υψηλό ποσοστό συμμετοχής, δηλαδή επιπέδων ή και καλύτερου επίπεδου από ό,τι διαπιστώνουμε στην Ευρώπη και ε, επίσης συμμετέχουν οι μειονότητες που παλιά θα μπορούσαμε να τις λέγαμε μειονότητες τώρα δεν είναι μειονότητες, είναι τμήμα του πολυεθνικού βολιβιανού κράτους η Σοφία Ευτυχώ, εκεί που οι Ινδιάνοι πήραν τι ζωέ του στα χέρια του και αποφάσισαν ποιο θέλει να του κυβερνάει και με ποιε πολιτικέ θέλουν να κυβερνιόνται. Κοιτάξτε, ποιοι μιλάνε για δημοκρατία σε, στην Ευρώπη. Ποιοι μιλάνε για δημοκρατία και σε ποια Ευρώπη μιλάμε για δημοκρατία. Και θα σα μιλήσω σαν Ελληνίδα αυτή τη στιγμή. Μιλάνε για δημοκρατία αυτοί που απείλησαν τον ελληνικό λαό ότι αν δεν ψηφίσει αυτόν που θέλουν εκείνοι, τα οικονομικά συμφέροντα κυρίω θα τιμωρηθεί ο ελληνικό λαό. Μιλάνε αυτοί που αλλάξαν την κυβέρνηση της Γαλλίας μέσα σε μια νύχτα. Μιλάνε αυτοί που κατεβάζουν κυβερνήσεις, μιλάνε για δημοκρατία, εκλεγμένες κυβερνήσεις από λαού, χωρίς να σέβονται τίποτα. Μιλάνε αυτοί που αλλάζουν εκλεγμένους πρωθυπουργούς με τραπεζίτες. Για ποια δημοκρατία μιλάνε. Αν δεν έχετε άλλες ερωτήσεις θα ολοκληρωθεί εδώ η μισή ώρα αυτής της συνέντευξης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν εδώ και όσους μας παρακολούθησαν από τα κομπιούτερ τους. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς.